το επόμενο σημείο. Πρόκειται για δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των ορών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης, ανάπαυσης. Έχει τον λόγο ο Επίτροπος κ. Μπαρό. Κύριε Πρόεδρε, θα σας διαβάσω την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των ορών οδήγησης και περιόδων ε, παύσεως ε, ο κανονισμός 261 του 2006 ίσχυσε από τις 11 Απριλίου 2007 δηλαδή εδώ και περίπου δύο χρόνια και αντικατέστησε τις ώρες οδηγήσεως και ώρες αναπαύσεως που δεν είχαν αλλάξει για μία εικοσαετία. Από όταν υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά την εφαρμογή του μέσω πολλών συνεδριάσεων με τα κράτη-μέλη, με τους ενδιαφερόμενους στην βιομηχανία, στα συνδικάτα και τις ομάδες εργασίας που έχουν δημιουργηθεί. Ή στο μέλλον η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το τη διετή έκθεση για την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων που δείχνει τι προσπάθειες έχουν γίνει από τα κράτη-μέλη αλλά διαπιστώνουμε ότι πρέπει να αυξηθούν για να φτάσουν στο επίπεδο το οποίο απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μεταξύ των ε, πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να αναφέρουμε τις καθευθυντήριες ε, γραμμές που δημοσιεύοντας κατόπιν στην ενέσω των κρατών μελών και αποβλέπουν στον ε, εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων ορών οδήγησης και επαύσεως εάν ο οδηγός χρειαστεί για ένα κατεπήγοντα λόγο να διακόψει την ανάπαξή του. Ε, επίσης η Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει τον ψηφιακό χρονοταχυγράφο διότι τον Ιανουάριο ε, ορισμένα μέτρα υιοθετήθηκαν για την βελτίωση του συστήματος και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταρτήσουν ειδικούς εξοπλισμούς για να παρακολουθήσουν και να ελέγχουν τους χρονοταχυγράφους. Ένα δεύτερο ε, σύνολο μέτρων για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών για τον χρονοταχυγράφο συζητείται στην επιτροπολογία. Μεταξύ άλλων τα μέτρα αυτά θα διευκολύνουν την ε, ε, χρήση του χρονοταχυγράφου ταχογράφου από τους οδηγούς απλοποιώντας τις καταγραφές διαχειρός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποβλέπει στη σωστή εφαρμογή του κανονισμού κατά τρόπον ώστε η, νέα εφαρμογή ε, να αποτελέσει ε, μία βελτίωση και γι' αυτό έπεισε η Επιτροπή της ε, χώρες που συμμετέχουν στην ΕΕΤΕΡ να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες από το 2010. Βεβαίως όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν οι κοινωνικοί κανόνες να εφαρμόζονται εναρμονισμένα στην Ευρώπη. Αυτά μπορούσα να πω στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ακούσω πολύ προσεκτικά τις παρεμβάσεις των διαφόρων Ευρωβουλευτών. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Για το ΕΛΚ, για δύο λεπτά, η κυρία Βόρτμαν Κόλ, παρακαλώ. Yeah, eh, Σας ευχαριστώ θερμά Σήμερα παρατηρείται κάποια σύγχυση ως προς αυτήν τη δήλωση της Επιτροπής, αλλά είναι προφανές ότι η προφορική ερώτηση του ΕΛΚ με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες είναι η βάση της συζήτησης που θα κάνουμε για αυτήν την δήλωση. Η προφορική ερώτηση λοιπόν προκύπτει από τις ανησυχίες που ακούγονται για την μεταφορά των κανόνων αυτών στην πράξη. Βλέπω ότι ας πούμε παράδειγμα ότι αν μετακινήσει κανείς το αυτοκίνητό του μπορεί να του επιβληθούν τρομερά πρόστιμα. Τι λέει. Και ιδίως η οδηγοί βαρέων οχημάτων μπορεί να παίρνουν πρόστιμα για μία απλή στάθμευση για διανυκτέρευση. Με χαρά άκουσα να λέτε ότι θα γίνει μια νέα έκθεση και ότι θα έχετε γνώση των προβλημάτων αυτών. Το θέμα δεν είναι να υπάρξουν απλώς καινούργιοι κανόνες, αλλά να εξετάσουμε πρώτα τους υπάρχοντες για να κάνουμε μια αξιολόγηση και να λάβουμε υπόψη μας τις συμβουλές που μας δίνουν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Η αξιολόγηση λοιπόν αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να ζητηθούν βελτιώσεις. Βέβαια όλα αυτά δεν έχουν ισχύ νόμου στα κράτη-μέλη και μπορεί τελικά να καταλήξουμε με άδεια τα χέρια αφού δεν είναι δεσμευτικές οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές. Ελπίζω εσείς κύριε Επίτροπε που γνωρίζετε το θέμα χαίρομαι ιδιαίτερα που αντικαθιστάτε τον κύριο Ταγιάννη θα κάνετε πραγματικά αυτή την αξιολόγηση. Ευχαριστούμε για, στη συνέχεια για τη Σοσιαλιστική Ομάδα κυρία Τικάου. Κύριε Πρόεδρε, ε, ο, κύριε Επίτροπε λαμβάνοντας υπόψη ε, το χρόνο οδηγήσεως και αναπαύσεως για τους οδηγούς και μεταφορείς, στις οδικές μεταφορές θα λάβει υπόψη και την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει ακόμη αρκετά μέτρα για να μειώσει τον αριθμό των οδικών ατυχημάτων. Βεβαίως θα πρέπει να βελτιωθεί από τα κράτη-μέλη ε, η εποπτεία και ο έλεγχος της κυκλοφορίας και θα ήθελα να αναλύσω την πρώτη έξερση Τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έπρεπε να είναι διετής αλλά άργησε να εκδοθεί και μέσω αυτής της εκθέσεως είναι προφανές ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν υπερβεί τον ελάχιστο ποσοστό των ελέγχων που έπρεπε να κάνουν και άλλα κράτη δεν, έφτασαν το, ε, δεν επέτυχαν το στόχο τους. Στην έκθεση Gross για την αγορά ε, συναντηθήκαμε με το Συμβούλιο και προσθέσαμε ένα συμβιβαστικό κείμενο το οποίο ζητά όλοι οι έλεγχοι της κυκλοφορίας να μην οδηγούν σε διακρίσεις αλλά ε, να λαμβάνουν υπόψη και το χώρο κατοικίας του μεταφορέα. Ε, να ξέρετε ότι μεταξύ της Ρωσίας και της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχουν ασφαλείς θέσεις ε, παρκαρίσματα αλλά όχι επαρκείς διότι 40% των ληστιών οι οποίες γίνονται από, ε, τους, επί των μεταφορέων γίνονται σε αυτές τις, τους χώρους σταθμέσεως. Ζητήσαμε λοιπόν να υπάρχουν ασφαλείς χώροι σταθμεύσεως και συγχρόνως να υπάρχει σεβασμός του χρόνου οδηγήσεως και αν υπάρχουν οι συνθήκες για τους οδηγούς. Για 1,5 λεπτό κυρία Λίχτενμπέργκερ παρακαλώ. herzlichen Dank. Σε ευχαριστώ θερμά Κύριε Πρόεδρε, η συνάδελφος από τη συντηρητική ομάδα είπε ότι ο τομέας έχει μεγάλες ανησυχίες. Αν για ένα λεπτό παραπάνω οδηγούν κάποιοι οι οδηγοί, εβδομάδες υστερότερα θα πρέπει να πληρώσουν βαριά πρόστιμα. Εγώ δυστυχώς υπό το δικό μου πρίσμα προσωπικά μπορώ να καθησυχάσω τη συνάδελφο για αυτό που εξέθεσε. Διότι είναι τέτοιου είδους οι έλεγχοι στα κράτη-μέλη χαλαροί και δεν υλοποιούν τα περισσότερα κράτη-μέλη τους ε, τα καθήκοντα ελέγχου που έχουν πλήρως ή αποδυναμωμένους ελέγχους ε, κάνουν και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στα σπάργανα ακόμα όσον αφορά τέτοιου είδους ελέγχους. Και αυτό παρότι έχουμε ολέθρια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όταν για παράδειγμα έναν ε, οδηγό τον σταματάει κάποιος σε ένα, σε ένα αυτοκινητόδρομο που επί 38 ώρες συνεχώς εργαζόταν, ε, τότε κανένας δεν μπορεί να πει ως δικαιολογία ότι δεν βρήκε ασφαλή χώρο στάθμευσης. Αλλά βλέπετε υπάρχει πίεση από πλευράς των εργοδοτών να οδηγούν οι οδηγοί τους μέχρι τελικής πτώσεως. Και αυτό είναι κίνδυνος για όλους τους άλλους που συμμετέχουν στι οδικέ μεταφορέ μεταφορές. Και για τα σοβαρά δυστυχήματα, ατυχήματα από πλευράς βαρέων ε, φορτηγών οχημάτων δεν χρειάζεται να πω εγώ το τι συμβαίνει, το ξέρουμε όλοι ότι είναι η κατάσταση καταστροφική. Και ιδιαίτερα όταν μεταφέρονται και επικίνδυνα αγαθά τα οποία σε τέτοια ατυχήματα προκαλούν και ζημιές, τεράστιες ζημιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν καλοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι έχουν ουσιώδη, θεμελιώδη σημασία εδώ. Δεύτερον, πιστεύω ότι ακριβώς στην εισαγωγή Υπότιτλοι AUTHORWAVE του ψηφιακού ταχογράφου, ναι μεν έχουμε μια μεγάλη ιστορία όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από τα κράτη-μέλη, επιτέλους όμως ήρθε η χρονική στιγμή, επιτέλους να καταστεί εφικτός και δυνατός καλύτερος έλεγχος. Καλύτερη έλεγχη προς όφελος των οδηγών, προς όφελος όλων όσων εμπλέκονται στις οδικές μεταφορές και στην κυκλοφορία και όλων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λίχτενμπεργκερ. Για 1,5 λεπτό για την ομάδα των ανεξαρτήτων δημοκρατών, ο κύριος Μπλόκλαν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτέλους η λειτουργία, η ρύθμιση των θεμάτων των ορών οδήγησης και ανάπαυσης έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν πάμπολα παράπονα για την μη ορθή εφαρμογή διατάξεων και πρέπει κάτι να κάνει κανείς. Πρέπει να επανεξεταστεί ταχύτατα ο κανονισμός. Τι πρέπει να γίνει καλύτερα. Η νομοθεσία. Η νομοθεσία πρέπει να είναι προβλέψιμη. Φυσικά δεν θέλω όλες οι ποινές και τα πρόστιμα να εναρμονιστούν. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είμαι υπέρ μιας ε, σαφούς ρύθμισης, προβλέψιμης ρύθμισης ε, και αντιμετώπισης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να παρεκκλίνουμε από μη ρεαλιστικές ποινές και πρόστιμα και από τις ε, από χρονοβόρες διαδικασίες. Τώρα, η σημερινή νομοθεσία κυρίως ε, για τους αλλοδαπούς οδηγούς ε, δημιουργεί τον κίνδυνο αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Αυτό δεν είναι θεμητό, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει. Είναι μια στρέβλωση της κοινής αγοράς, ε, της εσωτερικής αγοράς πρέπει να δει κανεί ε, το παράδειγμα ενό οδηγού. Κάποιο περνάει από τη Γαλλία και παίρνει, του επιβάλλεται ένα πρόστιμο επειδή δεν ε, ε, είχε επαρκή χρόνο ανάπαυση. Όμω, τι γίνεται σε σχέση με την ποινή, απαιτείται έξι ώρε εφαρμογή, ένα διάστημα έξι ωρών απαιτείται. Δεν μπορεί να οδηγήσει, να φορτώσει, να ξεφορτώσει ο οδηγό. Η πραγματική ζημιά λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερη από το πρόστιμο. Είναι πολλαπλάσια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε κύριε Επίτροπε, πρέπει σε τέτοιου είδους κράτη που δημιουργούν στρεβλώσεις για τον ανταγωνισμό να επιβάλλει κυρώσεις να μην δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Στρέφομαι προς τις χώρες του Νότου, αυτές εννοώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Περνάμε στο γύρο τώρα των άλλων αγοριτών Πρώτα απ' όλα για δύο λεπτά θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μαρινέσκου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Πρέπει να σεβόμαστε τις νενομισμένες ώρες οδήγησης και ανάπαυσης. Αυτό είναι ουσιώδες για να υπάρξει ασφάλεια στους αυτοκινητόδρομους και για τους οδηγούς και για τους επιβάτες Η Κομισιόν είχε ήδη προβλέψει μια σειρά μέτρων για τη χρησιμοποίηση του ταχογράφου και για να αυξηθεί ο έλεγχος από τα κράτη-μέλη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι μη οι οδηγίες και οι κανονισμοί για τις ώρες οδήγησης. Από τότε πρόκυψαν και νέα προβλήματα. Καταρχήν προβλήματα που αφορούσαν τον ψηφιακό ταχογράφο. Ψηφιακό ταχογράφο. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να σκεφτεί Πώς θα μεταφερθεί η οδηγία 22-2006 στην Εθνική Νομοθεσία των Κρατών Μελών και πώς με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού 561-2006 θα μπορέσει να προσαρμοστεί η Εθνική Νομοθεσία. Η Ρουμανία έχει εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της αλλά όχι μέχρι τέλους ακόμη ιδίως ως προς την εφαρμογή διαμεθοριακών κυρώσεων. Στη, κατά τη διετή έκθεση για τις χώρες μέλη ζητώ στην Κομισιόν να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει αυτό το θέμα του κανονισμού 561-2006. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό. Κύριος Λιμπεράτσκι, παρακαλώ. Panie Przewodniczący, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κάνουμε λόγο για τον χρόνο που αφορά την οδήγηση και ανάπαυση για τους οδηγούς ε, φορτηγών. Και συζητώντας αυτό το θέμα, μια και βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση, οι οδηγοί πλήττονται ιδιαίτερα από αυτή την κρίση επίσης και πολλές εταιρείε στον τομέα των οδικών μεταφορών δημιουργούν, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Το σημερινό σύστημα είναι περίπλοκο ούτως ή άλλως και δεν αποκλείει το να γίνονται σφάλματα το ζήτημα είναι να εφαρμόζονται οι κανόνες σωστά και δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις μέχρι σήμερα ότι λιγότερο αυστηροί κανόνες που θα επέτρεπαν την επέκταση του χρόνου οδήγησης ε, ανά εβδομάδα θα μπορούσαν να οδηγούν σε μεγαλύτερους κινδύνους ε, στους αυτοκινητοδρόμους μας. Από την άλλη πλευρά όμως αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και έχοντας όλο και μεγαλύτερες επιβαρύνσεις που δημιουργούνται για τους μεταφορείς στον τομέα των μεταφορών. Κάνουμε λόγο για την Ευρωβινιέτα εδώ και το, την εξωτερικοποίηση, το, την εσωτερική διαμόρφωση του εξωτερικού κόστου ε, δημιουργούν ε, ιδιαίτερα προβλήματα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα λάβει τον λόγο ο Επίτροπο Μπαρό, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Προφανώς άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία είπατε όλοι. Είναι προφανές ότι ο κανονισμός αυτός είναι σε μία περίοδο προσαρμογής. Ε, ροντάρουμε εφόσον μιλάμε για μεταφορές και είναι πολύ βασικό θέμα για την οδική ασφάλεια και για τον κοινωνικό τομέα. Θέλω λοιπόν να καθησυχάσω αυτούς οι οποίοι εξέφρασαν ε, ανησυχίες για το επάγγελμα διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει βαθμιαία να εφαρμοστεί ο κανονισμός ο οποίος έχει αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και είναι σε επαφή με τον κλάδο για την ερμηνεία του κανονισμού διότι υπάρχει τώρα και μία οδηγία η οποία καθορίζει τις συνθήκες των παραβάσεων και όσον αφορά τις ε, τα πρόστιμα θα προβούμε ε, σε μία έκθεση η οποία θα αποδείξει ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα μεταξύ κρατών μελών και ε, ταξινομούνται διαφορετικά και οι παραβάσεις. Επίσης θα ήθελα να σας πω και απαντώ εδώ στην κυρία Ρότμαν Κόλ η οποία αναφέρθηκε ή στην ανάγκη για τους οδηγούς να βρουν κάποιο πάρκινγκ, ε, πάρκινγκ ασφαλές. Η κυρία Ρότμαν Κόλ ε, ε, θυμάμαι ότι ή θέλατε να υπάρχουν περισσότεροι τέτοιοι ασφαλείς χώροι σταθμεύσεως και διότι πρέπει ίσως να οδηγήσει κανείς πιο πολλή ώρα για να βρει ένα τέτοιο ασφαλές χώρο στάθμευσης. Είναι σωστό κύριε Λιμπεράτσκι ε, όταν λέτε ότι δεν πρέπει να πιέσουμε πολύ το κλάδο αλλά ξέρετε κι εσείς ότι όλα αυτά γίνονται για να επιτρέψουμε να μην αναλυφθούν κίνδυνοι ασφάλειας και επίσης είναι κατά κάποιον τρόπο μια προστασία των οδηγών ενάντια σε ορισμένους κινδύνους που είναι έτοιμοι να αναλάβουν. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ μας ανέφερε τη σημασία των διατάξεων για την οδική ασφάλεια. Κύριε Μαρινέσκο, νομίζω ότι προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την εφαρμογή ε, σταθερά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ακόμη να συζητήσουμε τις ε, νομικές διατάξεις. Θα πρέπει να δώσουμε τον χρόνο, να συνηθίσουν όλοι και ε, θα είναι προς όφελος του τομέα εφόσον θα εναρμονίσουν καλύτερα τις συνθήκες εργασίας και από σεβασμό για την ζωή των οδηγών και επίσης για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτά είχα να σας πω. Βεβαίως ε, θα ε, διαμηνήσω στον φίλο μου ο Αντώνιο Ταγιάννη αυτά τα οποία είπατε για να προσέξει να συνεχιστεί αυτή η αξιολόγηση με στενή παρακολούθηση και ε, συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους και κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ για τα σχόλια που έγιναν απόψε από τους διάφορους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη τώρα είναι η συζήτηση <clears throat> για τη σύσταση για την δεύτερη ανάγνωση σε σχέση με την έκθεση της κυρίας Ντόιλ για τον καθορισμό <clears throat> ορίων καταλήπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Και θα δούμε τώρα αν η κυρία Ντόιλ δεν εμφανιστεί, τότε θα διακόψουμε τη συνεδρίαση για δύο λεπτά. Έτσι. Μέχρι ότου προσέλθει η κυρία Ντόιλ και εμφανιστεί στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ιδού κυρία Ντόιλ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ έγκαιρη και σκόπιμη η άφηξή σας. Δεν θέλω να την χαρακτηρίσω θριαμβευτική, αλλά είναι πραγματικά πολύ κατάλληλη η άφηξή σας. Είσαστε έτοιμοι να λάβετε τον λόγο κυρία Ντόιλ στα αγγλικά. You ready? Πολύ καλά. Εντάξει λοιπόν. Έχετε τον λόγο κυρία Ντόιλ. Όποτε είσαστε έτοιμοι μπορείτε να ξεκινήσετε. 10:30 και είχε προβλεφθεί. Είχα προσέξει ιδιαίτερα την ώρα στην οθόνη και δεν είναι ο Επίτροπος ο Επίτροπο Φερχόγγεν είναι καθοδόν. Εντάξει, να περιμένω ίσως, να προτιμώ να περιμένω δύο λεπτά μέχρι ότου να προσέλθει ο Επίτροπος Φερχόγγεν. Διότι ο Επίτροπος Φερχόγγεν και εγώ είχαμε επί δύο έτη διάλογο και συζήτηση για αυτή την έκθεση. Θα διακόψουμε για δύο λεπτά λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, μέχρι ότου αφηχθεί ο Επίτροπος Φερχόγγεν.